τρεις υποψήφοι ότι συμφωνούν με την πρόταση υποψηφιότητός τους. Η, η σύνθεση του Κοινοβουλίου σήμερα θα εμφανιστεί στα πρακτικά και